για ένα λεπτό, ενάμιση λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε. Καλώ ορίζονται στη συζήτηση αυτή και το ψήφισμα. Ελπίζω να υπάρχει ευρεία υποστήριξη από το Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό γιατί χρειαζόμαστε μια καλή εκκίνηση για το για τη διάσκεψη αυτή. Όχι μόνο εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά και πέρα από το Κοινοβούλιο κυρίω. Όντω η διάσκεψη θα πρέπει να επιφέρει αποτελέσματα και να βελτιώσει τα θεσμικά όργανα και τη λήψη αποφάσεων. Αλλά πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η διάσκεψη ελπίζω να δώσει απάντηση σε αυτό το έντονο αίσθημα που επικράτησε και μετά τις ευρωεκλογές όταν ήταν ρεκόρ οι πολίτε, ο αριθμό των πολιτών που ήρθαν να ψηφίσουν. Θα πρέπει να εμπιστευτούμε λοιπόν αυτό το αίσθημα των πολιτών για το μέλλον τη Ευρώπη. Θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή των πολιτών στη διάσκεψη. Είναι απαραίτητο αυτό και να δώσω μια σύντομη απάντηση στα σχόλια τη ακροδεξιά ότι πρόκειται να είναι μια διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη. Το άρθρο 19 είναι σαφέ. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ακούσουμε όλους στις υποψήφιες χώρες που θέλουν να συνεργαστούν μαζί μα. Είναι ευκαιρία αυτή η διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη να είναι μια διάσκεψη για μια πιο ισχυρή Ευρώπη σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Η ε, κυρία Μποναφέη, για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με τις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές οι πολίτες μας έδειξαν ότι θέλουν ακόμα να πιστέψουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ε, και ότι θέλουν να αλλάξει η Ευρώπη. Ε, οι κρίσεις που βλέπουμε γύρω από τα σύνορά μας είναι το τελευταίο καμπανάκι ε, κινδύνου και η τελευταία έκκληση για να αλλάξει η Ευρώπη. Οφείλουμε να ξεκινήσουμε με τη διάσκεψη αυτή ένα νέο στάδιο, μια νέα φάση μια δυνατότητα ε, να δοθεί ε, μια νέα πορεία στην Ευρώπη και ένας νέος ρόλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τρόπο ώστε να παθιάσουμε τους ε, πολίτες και να ακούσουμε προσεκτικά τις προσδοκίες τους. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια δυναμική και ορθολογική διάσκεψη η οποία θα είναι αξιόπιστη και αποτελεσματική. Αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε την ομφαλοσκόπηση αγαπητοί συνάδελφοι γιατί διαφορετικά αντί για ευκαιρία διάσκεψη θα γίνει στην ουσία καύσιμο ε, για τους αντιευρωπαϊστές, πράγμα που δεν θέλουμε. Κοιτάξτε, ε, λέει η Πρόεδρος, όταν ε, μιλούν οι ομιλητές τόσο γρήγορα, οι διερμηνείς έχουν πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Και όταν βλέπετε αυτό το φωτάκι της ταχύτητας, να μην πηγαίνετε ακόμα πιο γρήγορα, να επιβραδύνετε. Ε, κύριε Καμόν, ευχαριστώ. Η διάσκεψη της Ευρω... για την Εμπορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μια υπόσχεση. Μια υπόσχεση για την καλύτερη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαίρομαι που τα επόμενα δύο χρόνια θέλουμε να ρωτήσουμε τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι προστοκίες έχουν αυτοί για μια ισχυρή Ευρώπη στο μέλλον. Και το βασικό ερώτημα θα είναι το εξή. Ποιο είναι το δικό μας όραμα για την κοινή Ευρώπη. Και να ρωτήσουμε τους πολίτες ποιο είναι το δικό τους όραμα. Ε, αυτές οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις συχνά προκαλούν φόβο, φόβο τον οποίο δεν θέλουν να νιώσουν οι πολίτες. Αλλά η αίσθησή μου είναι ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ πιο θαραλέοι και τολμηροί από ό,τι φαντάζονται οι αρχηγοί κρατός και κυβερνήσεων. Και γι' αυτό λοιπόν αυτή την ε, τόλμη θέλουμε να την πάρουμε μαζί μας για να ληφθούν αποφάσεις για την καλύτερη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε πολλές προκλήσεις, όπως η καταστροφή του κλίματος. Πώς ε, να δώσουμε απαντήσεις αν δεν ε, ζούμε σε μια πιο ισχυρή και πιο ενωμένη Ευρώπη. Και πιστεύω ότι αυτή η διάσκεψη θα αποτελέσει και ε, μια ευκαιρία για να δώσουμε αυτό το πνεύμα για τα επόμενα χρόνια και γι' αυτό λοιπόν να υπάρξει αυτό το όραμα των ΗΠΑ της Ευρώπης. Ο κύριος Νίνας για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, μέχρι στιγμής ε, ακούσαμε από τη συζήτηση ότι έχουμε κρίση στην Ευρώπη. Και μάλιστα όχι μόνο μετά τι εκλογέ και πριν τι εκλογέ είδαμε ότι δύο πιθανότητε υπάρχουν. Λιγότερη ή περισσότερη Ευρώπη. Μέχρι στιγμή η ακροδεξιά εξέφρασε το δικό τη όραμα για το θέμα αυτό. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία θέλουν περισσότερη Ευρώπη και αυτή η πλειοψηφία κέρδισε τις εκλογές, η πλειοψηφία που θέλει περισσότερη Ευρώπη. Τώρα θα αποφασίσουμε πόσο περισσότερη Ευρώπη θέλουμε και αυτή την απάντηση θα πρέπει να τη δώσει το κοινό, οι πολίτες, να καθίσουμε όλοι να συζητήσουμε και να απαντήσουμε την ερώτηση. Η απάντηση στην ερώτηση μπορεί να είναι να θέλουμε λίγο λιγότερη Ευρώπη. Μπορεί αυτό να θέλει ο κόσμο. Λίγο λιγότερη Ευρώπη. Αλλά α αναλάβουμε αυτό το κίνδυνο. Γιατί μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι έχουμε καλύτερα επιχειρήματα. Γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη έφερε την ενότητα Ανατολής και Δύσης. Έχει φέρει ελευθερία, ειρήνη, ευημερία. Εμείς έχουμε πολλά εύστοχα επιχειρήματα και γνωρίζω ότι θα κερδίσουμε τη συζήτηση. Και μια και μιλάμε για συζήτηση. Ας συνεχίσουμε μια καλή συζήτηση στην Ολομέλεια και ας κάνουμε αυτή την πρώτη ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μπιτσότο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η Ευρώπη θα πρέπει να αλλάξει ε, από... να αλλάξει ολοκληρωτικά. Θέλουμε μια διαφορετική και νέα Ευρώπη. Ε, ε, αρκετά με την Ευρώπη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των τραπεζών, των, της γραφειοκρατίας. δεν θέλουμε την συνηθισμένη Ευρώπη του Μακρόν και της Μέρκελ. Θέλουμε την Ευρώπη των πτωχών, την Ευρώπη της πραγματικής δημοκρατίας και της ελευθερίας η Ευρώπη που θέλουμε να οικοδομήσουμε ε, πρέπει να σταματήσει την ε, παράτυπη μετανάστευση, ε, να προωθήσει το Made in Italy, να βοηθήσει να προστατέψει τους δικούς μας εργαζόμενους και τη βιομηχανία μας. Αυτή είναι η δημοκρατική Ευρώπη που θέλουμε και θέλουμε να την προχωρήσουμε με το κεφάλι ψηλά, με την πλάτη ίσια και με μεγάλη υπερηφάνεια. κυρία για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η ευγένεια, ο σεβασμός και η μετριοφροσύνη είναι χαρακτηριστικά των Βρετανών. Και εμείς συνεχίζουμε να είμαστε ένα έθνος που κρατάει τις υποσχέσεις του. Και όταν οι αξίες και αρχές μας απειλούνται, αρχίζουμε να αντιμαχόμαστε και να αντιπαλεύουμε αυτές τις στάσεις. Ε, ο Μπόρις Τζόνσον κέρδισε τις εκλογές. Ε, το Βρετανικό κοινό είδε ότι τρία χρόνια είχαμε καθυστερήσεις ε, και προδοσία ουσιαστικά της Βρετανικής Δημοκρατίας. Και όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του Brexit, θα πρέπει να μάθουμε κάποια διδάγματα για το μέλλον των σχέσεων μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η ιεραρχία κατάλαβε ότι δεν μπορεί πια να κοροϊδέψει το Βρετανικό λαό. Πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο για αποτελεσματική συνεργασία και φιλία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πάνω απ' όλα ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεχτεί επιτέλου την επιλογή των Βρετανών πολιτών να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ε, πολύ σωστά ανακεφαλαιώνει ο Βαλχάμσερ την κατάσταση όταν δυστυχώ έχετε ξεπεράσει το χρόνο σα, μιλάτε μόνοι σα Έχει διακοπεί το μικρόφωνο σα. οπότε σταματήστε, δεν έχει νόημα. Περνάμε στον επόμενο, στην επόμενη ομιλήτρια για 1,5 λεπτό, την κυρία Βόζεμπεργκ. κυρία πρόεδρε πριν τέσσερις μέρες δώδεκα νεκροί μετανάστες προσθέθηκαν στην τραγική λίστα θυμάτων μεταξύ τουρκίας και ελληνικών νησιών είκοσι άνθρωποι διασώθηκαν με υπεράνθρωπες προσπάθειες του ελληνικού ναυτικού ενώ δυστυχώς άλλοι τόσοι αγνοούνται. οι ροές μεταναστών συνεχίζονται αμύωτα παρά τις κακές καιρικές συνθήκες και η τουρκία εξακολουθεί κατά τη συνήθη πρακτική της να περιφρονεί το διεθνέ δίκαιο. το νέο σχέδιο ασύλου που έχει προμηνών εξαγγελθεί δεν έχει ακόμη προωθηθεί για ποιο μέλλον της ευρώπης συζητούμε σήμερα. δεν υπάρχει μέλλον χωρίς τη συμμετοχή όλων των χωρών στην αντιμετώπιση των κορυφαίων κοινών ευρωπαϊκών προβλημάτων. η έμφαση στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων που άλλωστε είναι μέλημα και κάθε κράτους μέλους σημαντική αλλά δεν αρκεί. απαιτείται δίκαιη και ίση κατανομή προσφύγων σε όλες ανεξαιρέτως τις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης με τα κριτήρια που έχουμε θέσει τίποτα δεν ακούσαμε σήμερα γι' αυτό. Πώ ονειρευόμαστε μια ενωμένη ευρώπη όταν κάθε κράτο μέλο ακολουθεί διαφορετική πολιτική ιδίων συμφερόντων όταν χώρε έχουν κλείσει τα σύνορα και αρνούνται να αναλάβουν ευθύνε, α είμαστε ρεαλιστέ και ειλικρινεί συνάδελφοι δεν μπορούμε να μιλάμε για το μέλλον μια Ευρώπη χωρί αλληλεγγύη στην πράξη. το μεταναστευτικό απειλεί τη συνοχή και τα θεμέλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η διαχείρισή του κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στι αξίε μας. έχουμε καθήκον και υποχρέωση να αντιδράσουμε άμεσα και έμπρακτα αλλά κυρίως σοβαρά και υπεύθυνα. σας ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μπάρλι για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερασπίσατε την ε, ειρήνη και την ασφάλεια στην ε, Ήπειρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμω δεν είναι τέλεια. Είναι μια διαδικασία ανεξέλιξη και αλλάζει διαρκώ. Θα πρέπει να γίνει πιο δημοκρατική, πιο οικολογική, πιο κοινωνική και κυρίω θα πρέπει να ξεπεράσει την απόσταση που νιώθουν πολλοί πολίτε προ αυτήν. Αυτό το, αυτή διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη είναι μια ευκαιρία. Αποφάσει ε, για του πολίτε ε, τη Ευρώπη που αισθάνονται ότι δεν εισακούονται. Θα πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Το καταλαβαίνουμε. Θέλουμε μια σαφή εντολή για τη διάσκεψη σε ό,τι αφορά τι πρωτοβουλίε και για την αλλαγή ενδεχομένω των συνθήκων. Είναι σημαντικό λοιπόν η διάσκεψη να έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και κατά δεύτερον, να συμμετέχουν οι πολίτε. Μόνο με τη σωστή επικοινωνία και με απόλυτη διαφάνεια μπορεί να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και αυτό είναι καθήκον του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Βόντεν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, εκατομμύρια πολίτε στη χώρα μα δεν καταλαβαίνουν καλά πώ λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούν ότι υπάρχουν μυθικοί κανόνε για τι μπανάνε, για διάφορα άλλα περίεργα πράγματα. Γιατί αυτό επικρατούσε επί δεκαετίε. Αλλά κοιτάξτε, δεν είμαστε οι μόνοι μα. Το Brexit είναι μια ένα παράδειγμα το οποίο θα μπορούσε να συμβεί σε πολλούς. Αυτό η διάσκεψη είναι ένα φιλόδοξο project και θα πρέπει να είναι φιλόδοξο αν θέλουμε να εξασφαλίσει το μέλλον της Ευρώπης των Εθνών. Πιστεύω ότι οι πολίτες θέλουν να αισθάνονται ότι εισακούονται και τους εκπροσωπούν. Εμείς ως οι ερετοί των πολιτών θα πρέπει να τονίσουμε ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει νομοθετική πρωτοβουλία για να αισθάνεται ο κόσμος ότι εισακούεται. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε αυτό. Και η μετανάστευση είναι ένα κλασικό παράδειγμα, γιατί οι εθνικέ κυβερνήσει μπλοκάρουν το Συμβούλιο. Η συνεργασία μεταξύ των λαών και των πολιτισμών και των κρατών είναι το μέλλον. Ο καθένα από μόνο του δεν μπορεί να αποτελέσει την απάντηση που δίνουμε στι προκλήσει του μέλλοντο. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Ντεπαρνέ, για ένα λεπτό. Και για μας τους πράσινους η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θέλει τα ερώτημα του πώς θέλουμε να ζήσουμε στο μέλλον. Τα οικολογικά, οικονομικά, κοινωνικά συμφέροντα, πώς θα διαμορφώσουμε. Αυτό μπορούμε το βρούμε μόνο αν ξεκινήσουμε μια μεγάλη αλλαγή απόψε με τους πολίτες. Η συμμετοχή είναι στο επίκεντρο μιας ε, βιώσιμης και ανανεώσιμης ε, κουλτούρας για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και της απώλειας της βιοπικιλότητας. Εδώ θα πρέπει να δούμε, για παράδειγμα, τι γίνεται με τη διατροφή μας. Πώς θα δημιουργήσουμε μια οικονομία, οικονομία αλλαγής για να μπορέσει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολλών. Αυτές οι διαδικασίες έχουν, ε, θα σημαίνουν βαθιέ τομέ και μπορούν να γίνουν μόνο αν υπάρχει δημοκρατική βάση ισχυρή. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι ιδιαίτερα που το Κοινοβούλιο σήμερα απευθύνει αυτή την πρόσκληση. Ελάτε να συμμετέχετε. Θέλουμε από κοινού να διαμορφώσουμε την Ευρώπη και θα πρέπει να προετοιμάσουμε την Ευρώπη για τι σημερινέ και μελλοντικέ προκλήσει. Τι Ευρώπη χρειαζόμαστε λοιπόν, Πώ θέλουμε να ζήσουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βιντεκομ, για ένα λεπτό. Η κυρία Γκαρσία Πέρες ε, μας θύμισε στην αρχή της συζήτησης ε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε με έξι χώρες ε, και το όραμα τότε ήταν να ε, ε, δημιουργηθεί μια συμμαχία χαλαρή ε, κυριάρχων κρατών με συνεργασία σε συγκεκριμένα θέματα και με την ευγενή ιδέα της προώθησης της ειρήνης. Και αυτή ήταν, αυτό, αν ήταν το όραμα ε, τότε ίσως ε, δεν θα έφευγε ε, τώρα η Βρετανία από αυτήν την ένωση. Όμως δημιουργήθηκε μία διαφορετική υπερκρατική δομή και πραγματικά εμείς θα είμαστε πάρα πολύ επιτυχημένοι στην κίνηση που κάναμε, την οποία ελπίζουμε να ακολουθήσουμε κι άλλοι. Και αν θέλουμε μέλλον για την Ευρώπη ή για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μάθετε το μάθημα, το δίδαγμα που σας διδάσκει το Ηνωμένο Βασίλειο. Συγγνώμη, δεν επιτρέπατε πια μπλε κάρτες. Σας ζήτησα συγγνώμη πριν, δεν έχουμε χρόνο. Κυρία Νίμπλερ, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Εκπρόσωπε του Συμβουλίου, κυρία Επιτροπή, αγαπητοί συνάδελφοι. Η διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη είναι σημαντική, γιατί όντω στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόμαστε να κάνουμε μεταρρυθμίσει σημαντικέ. Για μένα, ένα θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα τη ενίσχυση τη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Και όταν μιλάω για κοινοβουλευτική δημοκρατία, αυτό που εννοώ είναι η διαδικασία των κορυφαίων υποψηφίων, των Spitzenkandidaten. Καντιντάτων. Σήμερα, λοιπόν, μιλάμε για τους πολίτες. Εγώ διαπιστώνω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι από τις τελευταίες ευρωεκλογέ οι πολίτες έχουν χάσει μεγάλο το μήμα της εμπιστοσύνης της. Έχουμε πάνω από 200 εκατομμύρια ανθρώπους που συμμετείχαν στις ευρωεκλογέ. Και είχαν σαφείς προσδοκίες από εμά. Αυτοί που ψήφισαν ως ε, κορυφαίους υποψηφίου, στην τελική ανάλυση να είναι αυτοί που θα αναλάβουν την ευθύνη στην ε, Κομισιόν. Αν θέλουμε λοιπόν να κερδίσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών, θα πρέπει να προωθήσουμε τη μεταρρύθμιση της διαδικασίας των Spitzenkandidaten. Για, μας, για μένα η καρδιά της δημοκρατίας χτυπά εδώ στο Κοινοβούλιο. Εδώ λαμβάνονται οι αποφάσεις, εδώ χρειάζεται να συζητάμε και να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων. Είναι καλό να υπάρξει συμμετοχή των πολιτών προφανώς, αλλά στη τελική ανάλυση εμείς στο Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να αποφασίσουμε, γιατί γι' αυτό μα εκλέξανε. Και χαίρομαι Θα χαρώ αν ε, μέσα από τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης ενισχυθεί ακριβώς αυτή η θέση του Κοινοβουλίου στο κέντρο της Δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Ντόμπρεφ για ένα λεπτό. Ας είμαστε γενναίοι. Ας μιλούμε γενναία και θαραλέα. Ας αρχίσουμε να οικοδομούμε τα Ηνωμένα Έθνη της Ευρώπης. Έχουμε πετύχει πολλά τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά δεν αρκούν. Ο κόσμος αλλάζει, θα πρέπει και η Ευρώπη να αλλάξει. Οι απειλέ, οι προκλήσει αποκτούν παγκόσμιο χαρακτήρα. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει ένα παγκόσμιο παράγοντα. Και αντιλαμβάνομαι ότι ε, η προοπτική της αλλαγής φοβίζει, αλλά νομίζω ότι ο φόβος είναι κακό σύμβουλος. Γι' αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουμε και να δημιουργήσουμε μια πιο φεντεραλιστική, ισχυρότερη και δημοκρατικότερη Ευρώπη. Ας δημιουργήσουμε ένα συνασπισμό των γενναίων. Ας ε, δημιουργήσουμε τα, τις Ηνωμένε Πολιτείες, τα Ηνωμένα κράτη της Ευρώπης, ώστε οι επόμενες γενιές να είναι περήφανες για μας, όπως και εμείς είμαστε υπερήφανοι για τους ιδρυτές πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκινέα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, θέλουμε να εμπλέξουμε και τους πολίτες στη διαδικασία αυτή. Αλλά δεν θα πρέπει να είναι μόνο τυπική και για το Θεαθήνε αυτή η συμμετοχή. Υπάρχει τρόπος να εμπλέξουμε τους πολίτες ε, με τις συνελεύσεις των πολιτών ε, ή τις επιτροπές, τις κριτικές επιτροπές των πολιτών. Αυτή τη μέθοδο θα ήθελα να διαλέξουμε. Εγώ θα ήθελα, ε, Νίκολας, να είναι πρόεδρος της διάσκεψης ο Φερχόφστατ, γιατί χρειαζόμαστε μια ισχυρή ηγετική μορφή. Επίσης, ακόμη και συνάδελφοι από το κόμμα του Brexit που πολλοί θα μας λείψουν, τον άκουγαν με ιδιαίτερη προσοχή. Όλοι τον ακούγαμε με ιδιαίτερη προσοχή. Ας προωθήσουμε λοιπόν την υποψηφιότητα του Γκίφερ Χόφστατ ε, για να προεδρεύσει τη διάσκεψη, να ηγηθεί τις διαδικασίες για να έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση. Νομίζω όλοι περίμεναν με ανυπομονησία τη δική του κυρίως ομιλία. Ο κύριος Τόμπε. Μικρόφωνο παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, Κυρία Επίτροπε, τα προβλήματα της Ευρώπης δεν πρόκειται να επιληθούν με λιγότερη συνεργασία, αλλά αντίθετα με ενίσχυση της συνεργασίας και με τη δημιουργία μιας Ευρώπης που θα επικεντρώνεται στην αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα. Και είδατε πώς οργανωθήκαμε παντού στην Ευρώπη για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Θα πρέπει λοιπόν να μεριμνήσουμε ώστε να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη δημοκρατία και να αποφαινόμαστε με ενιαία φωνή σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Και αυτά τα θέματα θα τα πραγματευτεί η διάσκεψη της Ευρώπης. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για το εκλογικό σύστημα και για τις ε, θεσμικές αρμοδιότητες. Χρειαζόμαστε μία ε, ηγετική μορφή. Χρειαζόμαστε ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Μόνο έτσι θα προσετεριστούμε στην όλη διαδικασία και τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα πρέπει εμείς να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο, αλλά το περιεχόμενο του πλαισίου θα το δώσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες με τη συμμετοχή τους. Σας ευχαριστώ κύριος Μορένο Σάντσες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα ήταν ανέκαθεν ανοιχτό και διαφανέ σχέδιο που υπηρετεί το κοινό πεπρωμένο των Ευρωπαίων πολιτών. Δέκα χρόνια μετά τη θέση ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης Λισαβόνα, η διοργάνωση τη διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη θα μα δώσει μια μεγάλη ευκαιρία για να οικοδομήσουμε από κοινού με τους πολίτες το μέλλον τη Ευρώπη χάρη σε ένα συμμετοχικό και αντιπροσωπευτικό διάλογο σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Είναι πολλέ ιδέε που θα συζητήσουμε. Νομίζω όμω ότι ο πλήρη σεβασμό εκ μέρου του Συμβουλίου, τη διαδικασία του κορυφαίου υποψηφίου, το δικαίωμα νομοθετική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η εξάλληψη του δικαιώματο αρνησικυρία των μελών του Συμβουλίου και η μετάβαση στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία θα πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων. Ευελπιστώ ότι τα θεσμικά όργανα θα συνεργαστούν μεταξύ τους και με τους Ευρωπαίους πολίτες για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους επιδεικνύοντας πολιτική γενναιότητα κυρία Παγκάσαρ Ταντούρα. Ευχαριστώ. Είμαστε περισσότερα κάτι μέλη. Είμαστε κάτι περισσότερο από... Ε, δεν είμαστε όμως απομονωμένοι άνθρωποι. Υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις για όλους μας, οι οποίες δεν είναι εθνικές, είναι υπερεθνικές. Και αυτή είναι η ευκαιρία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα πρέπει να κοιτάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και να πορευόμαστε μαζί. Δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε, όμως, αν μας δηλητηριάσει το δηλητήριο του εθνικισμού. Φυσικά θα πρέπει να μάθουμε από, τον, από τις ακραίες τάσεις, από τον Brexit κτλ. Αλλά αν θέλουμε ένα μηχανισμό για να βαλκανοποιηθούμε, για να καταστρέψουμε την Ευρώπη, νομίζω ότι είναι κρίμα. Χρειαζόμαστε φυσικά να βάλουμε τους πολίτες στο κέντρο του συστήματος του ευρωπαϊκού συστήματος, του ευρωπαϊκού συστήματος. πρέπει η... να εξανθρωπιστεί η τεχνητή νοημοσύνη. Χρειαζόμαστε Ευρωπαίους πολίτες. Δεν πρέπει να καταστρέψουμε την Ευρώπη. Δεν πρέπει να πούμε ναι στα σύνορα. Ευχαριστώ. Σάιμον, 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, η ωραία συζήτηση έχει δείξει ότι 10 χρόνια μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας χρειάζεται μεταρρύθμιση των ε, συνθήκων. Ο υπέρτατο στόχος αυτή τη διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης θα έπρεπε να είναι η δυνατότητα διαπραγμότευσης των Ευρωπαίων να ενδυναμώσουν την Ένωση. Και επίσης είδαμε ότι σε μια τέτοια ωραία συζήτηση ε, δεν έχουμε μιλήσει για ε, το πώς ε, σε υπερεθνικό επίπεδο μπορούμε να οργανώσουμε το δημοκρατικό διάλογο. Είναι πολύ ωραία τα λόγια που ανταλλάσσουμε μεταξύ μας σήμερα. Μιλάμε για στοιχεία άμεση δημοκρατίας, κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Αλλά ένα πράγμα δεν πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να υπάρξει κανένας διαχωρισμός μεταξύ των όσων επιθυμούν οι πολίτες και το τι κάνει το κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο μπορεί να γίνει εξυπνότερο και πιο ενημερωμένο μέσω αυτή τη διάσκεψης, όμως με τα τελευταία τελευταία χρόνια μάθαμε στο Κοινοβούλιο ότι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι το καλύτερο μέσο για να οργανώσουμε το δημοκρατικό σύστημα. Ασχέτω από την έκβαση της διάσκεψης, θεωρώ σημαντικό για, το, ε, για τα ευρωπαϊκά κοινά να υπάρξει μια σωστή παρουσίαση και το Κοινοβούλιο να είναι πλατφόρμα για την εξέταση των ε, ευρωπαϊκών κοινών. Θα πρέπει λοιπόν εσεί. Πρόεδρε, να κοιτάξετε ότι και η συζήτηση, η Σύνοδο τη Ολομέλεια θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί. Δεν μπορεί από τη μια κάποιοι να αγορεύουν και από την άλλη κάποιοι απλώ να ε, παρίστανται. Θα πρέπει να δούμε πώ θα παρουσιάζονται οι διαπραγματεύσει και οι συζητήσει μα και στα μέσα μαζική ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ε, Ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό, ο κύριος Μπενιφέη. Η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης ε, είναι ένα φιλόδοξο project για διάλογο μεταξύ πολιτών και θεσμικών οργάνων, ούτω ώστε να προκύψει μια πρόταση μεταρρύθμισης για την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση συγκεκριμένους στόχους. Θα πρέπει να προσέξουμε το περιεχόμενο και να δώσουμε στην Ευρώπη τη δυνατότητα να ασχοληθεί με αυτά ε, πάνω σε θέματα που επηρεάζουν πολύ τη ζωή μας την φορολογία, την καταπολέμηση κλιματική αλλαγή, τι κοινωνικέ πολιτικέ, η εξωτερική πολιτική, που μας ενδιαφέρει και είναι πολύ επίκαιρο θέμα τελευταία. Θα πρέπει τα συμπεράσματα της ε, διάσκεψης να γίνουν σεβαστά, να υπάρξει συνέχεια μέσω συγκεκριμένων νομοθετικών μέτρων, μέσω της ε, τροποποίησης των συνθήκων. Χρειαζόμαστε την, ε, μια ομοσπονδία. Με αυτό θα έχουμε τον καλύτερο θα έχουμε τα καλύτερα εχέγγυα ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε τη διάσκεψη ως πολιτική βετρίνα για να κατεβάσουμε τον πύχη. Θα πρέπει να το εμποδίσουμε αυτό για το καλό της Ευρώπης, για το μέλλον της Ευρώπης. Μπουαγέ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, όλοι βλέπουμε στο κοινοβούλιο αυτό, η βασική πρόκληση είναι να δούμε πώ θα λειτουργούμε εμεί εσωτερικώ. Και πολλέ φορέ δυσκολευόμαστε ε, για να καλύψουμε το χάσμα μεταξύ αυτού που αισθάνονται οι Ευρωπαίοι πολίτε και καταλαβαίνουν για τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Κοινό μα στόχο, κοινό στόχο αυτή τη διάσκεψη θα πρέπει να είναι να αποσαφινιστεί ο τρόπο λειτουργία μα και ξεκινάμε από την σαφήνεια την πλέον καθοριστική στιγμή, τη στιγμή των ευρωεκλογών. Τότε πρέπει οι πολίτε που είναι ευαισθητοποιημένοι να καταλαβαίνουν τι γίνεται. Ε, τον περασμένο Μάιο ο μηχανισμό των κορυφαίων υποψηφίων φάνηκε ω μια πρακτική λύση, αλλά έδειξε ότι δεν λειτουργεί. σα ίσα θα είναι πιο σκόπιμο αν ταυτόχρονα οι Ευρωπαίοι πολίτε μπορούν να αποφανθούν για τι ε, υπερεθνικέ, για του υπερεθνικού ε, υποψηφίου και του εκλογικού τα Τα ευρωπαϊκά ψηφοδέλτια για τις ευρωπαϊκές εκλογές νομίζω ότι είναι ο καλύτερος στόχος. Ευχαριστούμε ο κύριος Ρέσλερ για 1,5 λεπτό. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα διαφέρει σημαντικά από ε, πριν από μία δεκαετία όταν τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Βλέπουμε άνευ προηγουμένου τεχνολογικές, οικονομικές αλλά και δημογραφικές αλλαγές. Αυτό σαφώ επηρεάζει τη ζωή μας, τον τρόπο που εργαζόμαστε και τον τρόπο που επικοινωνούμε. Έχει όμως και αντίκτυπο στην ε, πιο ε, ενεργό συμμετοχή των πολιτών ε, στη δημοκρατία μας. Γι' αυτό είναι ευθύνη μας να προσφέρουμε νέους και καινοτόμους τρόπους στους Ευρωπαίους ώστε να συμμετέχουν περισσότερο στις αποφάσεις που τους αφορούν. Οι νέοι Ευρωπαίοι συχνά ε, βρίσκονται επικεφαλής ε, στις μεταρρυθμιστικές τάσεις των κοινωνιών μας ε, και μπορούν να προσφέρουν μια νέα οπτική. Χαίρομαι που η Αντιπρόεδρο Σουίτσα θα ηγηθεί των εργασιών της διάσκεψης, διότι είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε όλη την ποικιλομορφία της Ευρώπης, να συμπεριλάβουμε όλες τις ιδιαίτερες οπτικές των πολιτών από όλες τις γωνιές της Ευρώπης και για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να συμπεριλάβουμε όλες αυτές τις πτυχές. Η διάσκεψη αυτή ε, δεν ε, θα πρέπει να είναι μια άσκηση ρουτίνας, ε, θα πρέπει να εργαστούμε επικοδομητικά, συμμετοχικά και να προσαρμόσουμε την Ευρώπη στο νέο κόσμο και για τις νέες γενιές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φρίτσο. Ένα λεπτό. I'm Oh, oh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, κυρία ε, Πρόεδρε και κυρία Πίτροπε. Οι δημοκρατικές αξίες, η αλλαγή του κλίματος, ε, η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισότητα είναι τα σημαντικά θέματα που ε, θα πρέπει να καλύψει η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Μία διάσκεψη που θα πρέπει να απευθυνθεί και στις νεότερες γενιές. Χαίρομαι εδώ σήμερα που άκουσα μια ζωντανή συζήτηση όπου πολλοί από τους νέους ε, και νεοεκλεγέντες ε, βουλευτές έχουν αναλάβει πρωτοβουλία στην συζήτηση αυτή. Η συζήτηση για το μέλλον θα πρέπει να έχει θέμα τα ε, θέματα που ενώνουν και που ενισχύουν την Ευρώπη. Θα πρέπει να υπερασπιστούμε την Ευρώπη, θα πρέπει να δώσουμε ελπίδα στη νέα γενιά για το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, κύριο Στροτσάνη. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ευκαιρία να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Μπορούμε να δώσουμε νέα ορμή στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική. Η συμμετοχική δημοκρατία είναι σημαντική, θα πρέπει όμως να φροντίσουμε ε, να ε, ε, μην ε, επιβάλλουμε σε άλλους την ιδεολογία μας. Ε, ε, είναι σημαντικές οι παραδόσεις αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της Ευρώπης. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τις παραδοσιακές μας αξίες, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε τι είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής. Η ευρωπαϊκή ταυτότητα ε, μπορεί να προστατευτεί μόνο εάν προστατεύσουμε και τις αξίες των εθνικών κρατών. Θα πρέπει να θεωρήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ένωση αξιών όπου υπάρχει ποικιλομορφία, η οποία όμως βασίζεται στα ε, εθνικά κράτη. Γι' αυτό δεν μπορούμε να δεχτούμε τις Ηνωμένε Πολιτείες της Ευρώπης. Ο κύριος Τιμόσεβης, για ένα λεπτό. Η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης έρχεται στην καλύτερη χρονική στιγμή. Το, τα τελευταία 25 χρόνια άλλαξε η κοινωνία. Ε, έχουμε καινούργιες τεχνολογίες, ε, η Δημογραφική έκρηξη σε πολλέ περιοχέ, ε, κλιματική κρίση. Γι' αυτό πρέπει να δράσουμε. Η Ευρώπη πρέπει να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα και οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να καταλάβουν την ε, νέα κατάσταση. Η διάσκεψη πρέπει και μπορεί να διαγνώσει τα προβλήματα και να δώσει συνταγέ και λύσει. Η προπόθεση για την επιτυχία είναι η άνευ συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών Διαβουλευσει, διασκέψεις, όλα αυτά χρειάζονται, αλλά δεν είναι απαραίτητα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πλήρω την ε, επιγραμμική επικοινωνία. Ο καλύτερος τρόπος είναι να έχουμε πανευρωπαϊκά συμβουλευτικά δημοψηφίσματα με συμμετοχή εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτό είναι δημοκρατία. Οι πολίτε θα αισθανθούν ενεργοί και θα αισθανθούν ικανοποίηση επειδή θα πούν την άποψή του. Μαϊντέλ, για λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αντιπρόεδρε, η ιδέα του να έρθουμε σε επαφή με τους πολίτες μας είναι βασικό εργαλείο, δεν είναι ψυχαγωγία. Θα πρέπει να ρωτήσουμε τους ε, πολίτες μας πώς βλέπουν την Ευρώπη με ειλικρίνεια και τιμιότητα και επικοδομητικά. Εάν λέμε ότι πρέπει να τους ακούσουμε, θα πρέπει να είμαστε και έτοιμοι να λάβουμε υπόψη αυτά που θα πούν και να τα εφαρμόσουμε. Θα είναι η μεγαλύτερη άσκηση άμεση δημοκρατία στην Ευρώπη τις τελευταίες ε, δεκαετίες και δεν θα πρέπει να έχουμε έτοιμε ήδη λύσει. Ε, σε ορισμένε πρωτεύουσε ετοιμάζονται και ομιλίες και νέες συνθήκες ε, και νέα μπλοκαρίσματα, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τι λέει ο κόσμος. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα θελήσει απλώς να πει το ok χωρίς να μιλήσει ουσιαστικά. Το θέμα δεν είναι να έχουμε αφήσει και να επινοήσουμε μηχανισμούς για να καθοδηγήσουμε τη δημόσια συζήτηση. Θα πρέπει να ακούσουμε και να εφαρμόσουμε αυτά που θα μας πούν. Αυτές οι κακές συνήθειες, οι παλιές συνήθειες, είναι ακριβώς ο λόγος γιατί θα πρέπει να έρθουμε εκ νέου σε επαφή με τους πολίτες μας. Ο κύριος Γκλουξμαν, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ε, επί πολλά χρόνια τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είχαν την ε, ιδέα ότι μπορούν να φτιάξουν την Ευρώπη χωρίς τους ε, ανθρώπους. Για τους ανθρώπους, αλλά χωρίς αυτούς. Όχι εναντίον τους, αυτά τα λένε οι ακραίοι. Αλλά σήμερα φτάσαμε στην άκρη της Αβίσου. Ναι, αυτή η διάσκεψη για να επαναδημιουργήσουμε την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκ των όνου Αλλά θα πρέπει η συζήτηση να φύγει από τους θεσμούς και να τροφοδοτήσει ολόκληρη την κοινωνία, πώς θα φτιάξουμε κοινό στρατό, ε, πώς θα έχουμε κοινή φορολογία. Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα θα πρέπει να συζητηθούν και να αποφασίσουν πάνω σε αυτά με τους περισσότερους πολίτες στο πλευρό μας. Δεν πρέπει απλώς να διαβουλευτούμε, αλλά να χτίσουμε μαζί. Θα πρέπει να είναι μια νέα αρχή αυτή, όχι μόνο λόγω των συμπερασμάτων, αλλά και λόγω της μεθόδου. Θα πρέπει να δημιουργηθεί πραγματικά ένας ενεργός και όχι παθητικό Ευρωπαίος πολίτης, να γίνει μια υπερεθνική δημόσια συζήτηση. Είτε θα εκδημοκρατιστούμε ή θα πεθάνουμε. Ε, τι προτιμούμε, τον εκδημοκρατισμό. Ο κύριο Μπούντα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το μέλλον της Ευρώπης είναι αναμφίβολα μια μέρημνα μεγάλη σημασία για όλους μας. Και κερδίζω την πρωτοβουλία αυτή να ξεκινήσουμε σήμερα να θέτουμε τα θεμέλια για το μέλλον τη Ευρώπη μέσω αυτή τη διάσκεψη. Θα είναι μια ευκαιρία οι πολίτε να μπορούν να εκφράσουν τι απόψει του, τα δικά του ε, θέλω για το μέλλον τη Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό να δεχτούμε τι συνεισφορέ των πολιτών στην οικοδόμηση του μέλλοντο τη Ευρώπη. Ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνονται σεβαστέ οι αναλύωτες και απαλωτρίωτες αρχές μας. Θέλουμε μια Ευρώπη που να προστατεύει το κλίμα, το περιβάλλον, τα κοινωνικά δικαιώματα, την εργασία. Για όλα αυτά χρειάζονται εχέγγυα. Και βεβαίω όλα θα καθοριστούν από τι τελικέ αποφάσει. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε ένα βήμα στου πολίτε για να μπορούν να εκφράσουν τι απόψει του και να μα προτείνουν λύσει για αυτό που θεωρούν σωστό για μια εύρωστη Ευρώπη. Ευχαριστούμε κυρία Κομπούλα Νάτρη για ένα λεπτό. Πρόεδρε, το κοινοβούλιο εδώ, τουλάχιστον η μεγάλη πλειοψηφία, είναι ανοιχτό, είναι ανοιχτό και έτοιμο για το μέλλον της Ευρώπης και όχι στα παρασκήνια. Ε, εδώ θέλουμε οι πολίτες να συμμετέχουν σε μία ε, ε, αγορά σαν την Αθηναϊκή για να μπορούν να λάβουν το λόγο, ιδίω οι νέοι, και να πούν τι θέλουν για το μέλλον της Ευρώπης. Το είδαμε με τη συμμετοχή των ευρωεκλογών του περασμένου Μαΐου. Αυξήθηκε κατά 12% η συμμετοχή τουλάχιστον των νέων. Τι θέλουμε λοιπόν για το μέλλον. Οι χώρε οι σκανδιναβικέ θέλουν εξωτερική πολιτική ασφάλεια, ίσε εργασιακέ ευκαιρίε και η Ευρώπη να αναλάβει έναν ισχυρότερο πρωταγωνιστικό ρόλο. Έχουμε αναλάβει δράση για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Θέλουμε κοινωνική δικαιοσύνη να πάψει το φιλετικό μίσο και η φορολογική απάτη. Θέλουμε η Θέλουν οι πολίτε να διευκολυνθεί η καθημερινότητά του και η διαβίωσή του, όμω η έλλειψη νομοθεσία δυσκολεύει πολλά πράγματα. Είναι πολλά λοιπόν τα θέματα που ανακύπτουν πάντοτε αμέσω πριν τι εκλογέ. Η διάσκεψη αυτή πρέπει να ασχοληθεί με το δημοκρατικό μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το σύστημα των κορυφαίων υποψηφίων, των speech and candidate, πρέπει να αποσαφινιστεί μέχρι τι επόμενε εκλογέ. Ευχαριστούμε ο κύριο Ντιτιέ για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα είναι ακόμη ε, ένα στοιχείο για να μπορέσει ο Εμμανουέλ Μακρόν να προετοιμάσει την ε, επόμενη προκλητική του εκστρατεία ή θα ωφελήσει πραγματικά του λαού. Θα το δείξει το μέλλον. Εάν θέλετε όμω συγκεκριμένα βήματα, να μια πρόταση. Ε, ξελέγημε στι 26 Μαου. Η θητεία μα διαρκεί 5 έτη. Ωστόσο, η πραγματική πραγματικά διαρθρωτική δουλειά μα ξεκινάει μόλι αυτή την εβδομάδα, δηλαδή 8 μήνε μετά την εκλογή μα. Πόσο χρόνο χάσαμε μέχρι να καταφέρουν να αναλάβουν τα καθήκοντά του τα διάφορα θεσμικά όργανα. Για τη διάσκεψη του μέλλοντο τη Ευρώπη, λοιπόν, προτείνω πολύ ε, συγκεκριμένα από την επόμενη θητεία το Συμβούλιο για ε, το και η Επιτροπή ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλαμβάνουν τέσσερι εβδομάδε μετά από τι ευρωεκλογέ το αργότερο και να ξεκινάνε όλα την 1η Ιουλίου και όχι την 1η ε, Ιανουαρίου του ερχόμενου έτου. Να μπορούν τα θεσμικά όργανα να λειτουργούν πλήρω και να ξεκινάνε τη δουλειά του ε, για το όφελος ε, για το καλό των λαών. Δεν μας έχουν εκλέξει για να παίξουμε τα πολιτικά μας παιχνίδια εδώ κυρίε και κύριοι, αλλά για να ετοιμάσουμε το μέλλον των λαών τη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα προχωρήσουμε στη διαδικασία Catch the Eye. Απλά θα ήθελα να πω ότι θα είμαστε πολύ αυστηροί όσον αφορά το χρόνο και θα παρακαλέσουμε και το Συμβούλιο και την Κομισιόν να, να καταλάβουν ότι έχουμε επίσημη ε, συνεδρίαση στι 12 και αυτό πρέπει να κλείσουμε παρά 5. Ο κύριο Κάνιεφ, ένα λεπτό ακριβώ έχετε στη διάθεσή σα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, σήμερα αποφάσισα να μιλήσω στα γαλλικά. Γιατί θέλω να εκφράσω την αγανάκτησή μου κατά τη ιδέα μια Ευρώπη πολλαπλών ταχυτήτων. Αυτήν ανέφερε ο πρόεδρο Μακρόν και είναι ο βασικό υποστηρικτή τη. Η Ευρώπη μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικέ πορείε, διαφορετικέ ταχύτητε για κάποια θέματα αυτό όμω βολεύει κυρίω του γραφειοκράτε και τι διοικητικέ υπηρεσίε. Ταυτόχρονα και ωστόσο η συζήτησή μα δεν ε, αφορά το καλό των κυβερνήσεων. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο καλό και το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, εκείνοι φτιάχνουν την Ευρώπη. Οι χώρε επίση που συνεργάζονται μαζί μα, όπω η Βόρεια Μακεδονία ή η Αλβανία. Το μέλλον δεν μπορεί να χτιστεί με διαφορετικέ ταχύτητε όταν οι χώρε θέλουν να επιτύχουν ευημερία, κράτο δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα. Το να έχουμε μια Ευρώπη με διαστρωματώσει και κατηγοριοποιήσει είναι πολιτικό σφάλμα και θα έχει ε, παρενέργειε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριο Λόπε Αγγιλάρ. Πρόεδρε, το 2009 τελικά μετά από πολλή προσπάθεια μπήκε τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Ο Φαν Ρομπάι ανακοίνωσε εδώ θα ήταν είπε ότι η Λισαβόνα, η συνθήκη τη Λισαβόνας θα ήταν η συνθήκη με την οποία θα ζούσαμε όλη μας τη ζωή. Και όμως η Ursula von der Leyen δρομολογεί μία διάσκεψη για την Ευρώπη που θα οδηγήσει και στην ε, αναθεώρηση τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Με τη Λισαβόνα είχαμε φοβερέ ανισότητε. Ε, το άρθρο 7 για εναντίον δύο κρατών μελών, ένα κρατος μέλος που φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλο και περισσότερα έδρανα εδώ που εκπροσωπούν ε, υπερεθ, υπερεθνικιστές, ε, ακραίους, ε, αντιδραστικούς και τελικά εμείς είμαστε το μοναδικό όργανο το οποίο είμαστε εκπροσωπευτικό. Έχουμε νομοθετική εξουσία, έχουμε νομιμότητα, αλλά θα πρέπει να υποφεληθούμε από την ευκαιρία που έχουμε με την διάσκεψη για να έρθουμε σε επαφή με τους πολίτες. Επόμενος ομιλητής, κύριος Φλέγκο, για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης αποτελεί ε, καταπληκτική ευκαιρία για να ακούσουμε τι ακριβώς θέλουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Τι σημαντικό είναι να ακούσουμε τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους και με τον τρόπο αυτό να δούμε πώς μπορούμε να μεταρρυθμίσουμε την Ευρώπη. Το κρίσιμο θέμα είναι πώς να ε, μετρήσουμε την επιτυχία της διάσκεψης με δύο τρόπους. Πρώτον, με βάση τα συμπεράσματα που θα πρέπει να υλοποιηθούν και δεύτερον, ε, ε, ανάλογα με τον αριθμό των πολιτών που θα συμμετάσχουν στη διάσκεψη. Γι' αυτό σημαντικό είναι να κινητοποιήσουμε τους πολίτες να συμμετάσχουν να ε, του αποζημιώσουμε για τα έξοδα μετακίνηση ε, και να φροντίσουμε να συμμετάσχουν μη κυβερνητικέ οργανώσει και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς ε, και όχι να ρωτάμε τους πολίτες μόνο μία φορά στα πέντε χρόνια πώ θα ήθελαν να είναι η Ευρώπη. Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια να τους δώσουμε την ευκαιρία να μιλήσουν. Ευχαριστώ κύριε Ζωτζίνσκι. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι ήδη από την αρχή της συζήτησης αυτής στις 9 η ώρα ήμουν εδώ και άκουσα όλους τους ομιλητές. Σέβομαι όλες τις απόψεις. Μερικές μπορεί να μου φάνηκαν περίεργες, αλλά θα ήθελα να απευθυνθώ στην αριστερά του ημικυκλίου. Είπατε πόσο σημαντική είναι η φωνή των Ευρωπαίων πολιτών. Ποια είναι τα γεγονότα όμως. Ε, Αυτή που έλαβαν τους περισσότερους ψήφους, όπως η πρώην Πρωθυπουργός μας, δεν εξελέγει πρόεδρος της, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από το ECR δεν εξελέγει ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου λόγω των δικών σας ψήφων. Ε, λέτε λοιπόν ότι θα έχουμε τη διαδικασία του Spitzenkandidat, ποια είναι τελικά η θέση του κυρίου Φερχόφστατ και θα πρέπει να θυμίσουμε αυτό που είπε ένας από τους πατέρες της Ευρώπης. Και κλείνει το μικρόφωνο. Ένα λεπτό ομιλίας έχετε μόνο, λέει πρόεδρος. Ο κύριος Μποτένκα, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι εδώ στα δεξιά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν πολύ εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιοι σοσιαλιστές και κάποιοι πράσινοι. είχαμε ανθρώπους προσέλευση των πολιτών στις εκλογές, ε, αλλά παρόλα αυτά έχουμε μια κρίση, γιατί οι ε, Γάλλοι και οι... Οι Ολλανδοί καταψήφισαν ε, το ε, Σύνταγμα, η Ιρλανδία καταψήφισε την ε, συνθήκη της Λισαβόνας, οι Έλληνες καταψήφισαν το μνημόνιο, αλλά δεν θα λυθεί η κρίση με μια διάσκεψη στην οποία να, να συμμετέχει μόνο η ελίτ υπό τον Γκίφερ Χόφστατ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Επίτροπο Σουίτσα, πρώην συνάδελφο. Ευχαριστώ. Dear President, honorable members, first of all, let me thank you for this uh, very vivid... Πρόεδρε, συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, ζωντανή συζήτηση που είχαμε. Λαμβάνω γνώση των απόψεών σας. Ε, ρόλος μου άλλωστε είναι να ακούσω τις απόψεις σας. Εναρκτήρια ε, ημερομηνία της διάσκεψης θα επιβεβαιωθεί, αλλά ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία, οι συνομιλίες και ήδη έχουμε συνομιλίες με όσο γίνεται περισσότερους παράγοντες. Τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη ήδη κάνουν ό,τι μπορούν για να φέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στου πολίτε. Ε, τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειε και να θυμόμαστε πώς αυτά συνδέονται με άλλους τομείς το, της αρμοδιότητάς μου, διότι είμαι αντιπρόεδρος ε, για την δημοκρατία. Θέλουμε λοιπόν να ακούσουμε τις απόψεις ανθρώπων όλων των ηλικιών. Θέλουμε να ακούσουμε και τους νέους. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την σημερινή συζήτηση. ήθελα να ευχαριστήσω τον Ντάνιελ Τουράντ ε, και όσους άλλους ανέφεραν τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Φυσικά δεν ξεχάσαμε τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ε, αρχική μας, ε, ήδη από την αρχή η ιδέα μας ήταν να συμμετάσχουν. Θα πρέπει να σκεφτούμε και τις μεγαλύτερες ηλικίε, διότι θέλουμε να συμβάλλουν ενεργά στην κοινωνία και την οικονομία μας όχι μόνο μη κυβερνητικέ οργανώσει ε, και οι πιο ηλικιωμένοι, αλλά και οι μειονότητε και φοιτητέ θέλουμε να συμμετάσχουν, ε, όπω και τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ, δήμαρχοι. Ε, Όποιο έχει να πει κάτι για τα θέματα που θα καλύψει η διάσκεψη. Οι απόψεις ε, αυτές ε, θα αποτελέσουν τη βάση για τις εργασίες μου ε, για την δημοκρατία. Η δημοκρατία μας χρειάζεται δημιουργικές και καινοτόμες λύσεις. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής, όποια και να είναι, θα πρέπει να είναι αυτά, θα πρέπει να υλοποιηθούν και θα πρέπει να βασίζονται σε αυτά που θα ακούσουμε από τους πολίτες μας. Όπως είπα ήδη, ε, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε πια τη ρουτίνα. Θα πρέπει να προσεγγίσουμε τη διαδικασία αυτή με καινοτόμο τρόπο και δημιουργικό. Ε, θέλουμε να έχουμε πλήρη συμμετοχή των πολιτών ε, και διαζώσεις και από το διαδίκτυο. Θα φροντίσω να ακουστεί η κάθε φωνή, να αφουγκραστούμε όλες τις φωνές και να δοθεί η κατάλληλη συνέχεια. Δεν θέλω να προδικάσω αυτά που έχουν να πούν οι πολίτες. Αντιθέτως, θα ήθελα να με εκπλήξουν. Και είμαι βέβαιη ότι και εμείς θα μπορέσουμε να εκπλήξουμε τους πολίτες ε, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να το πετύχουν αυτό μόνο εάν συνεργαστούμε στενά ως πραγματική εταίρη, Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστούμε, κυρία Σουίτσα. Και τώρα ο υπουργό Γκαντζάκ. Ή υπουργό Γκαντζάκ. Κυρίε και κύριοι, κύριοι βουλευτές, κυρία Σβίτσα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Άκουσα προσεκτικά τις θέσει του Ευρωκοινοβούλου ε, και τις απόψεις για τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Η διαδικασία αυτή απαιτεί ένα μακρόπνο όραμα και θα πρέπει να επικεντρωθούμε στους πολιτικούς στόχους που θα απασχολούν ε, πάνω απ' όλα τους πολίτες μας για τα ερχόμενα χρόνια. Ε, να, να σας διαβεβαιώσω ότι από την πλευρά της ε, δικής μας Προεδρίας θα φροντίσουμε να, να ε, αποσαφινιστεί και η θέση του Συμβουλίου για τα θέματα αυτά σε συνεργασία πάντοτε με το σώμα σας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως υπόθηκε ο Πρόεδρος σας όλοι και Αντιπρόεδρος Σουίτσα, ε, με τη συνεργασία όλων θα φροντίσουν να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις ιδέες σας. Και είμαι βεβαίω ότι μπορούμε να υπολογίζουμε στην εμπιστοσύνη σας για να βρούμε την κατάλληλη μορφή ώστε η πρωτοβουλία αυτή να ξεκινήσει με κοινέ βάσεις και να φέρει χειροπιαστά αποτελέσματα για τους πολίτες μας ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε ε, για την ταχύτητα και την ε, σαφήνεια. Ε, έχουμε λάβει προτάσεις ψηφισμάτων για τη συζήτηση αυτή. Έχει λήξει η συζήτηση. Θα ψηφίσουμε τα ψηφίσματα αργότερα σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ έντονη και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Προτού έχουμε την πανηγυρική μας συνεδρία. E ο πρόεδρο και αυτό εξοχότητα ο πρόεδρο Αμπουλά 2 τη Ιορδανία. Abbiamo Καλησπέρα σας συνάδελφοι. Έχουμε την τιμή να έχουμε σήμερα μαζί μας στην Ολομέλεια την αυτού μεγαλειότητα των βασιλιά Απτάλα 2 της Ιορδανίας, του Χασαμετικού Βασιλείου της Ιορδανίας. Είναι μεγάλη τιμή για μας. Επιστρέφει στο Ευρωκοινοβούλιο είχε προσκληθεί ξανά στο Κοινοβούλιο πριν από κάποια χρόνια. Ε, θα του δώσω το λόγο για την ε, ομιλία του. Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, φίλοι, σας ευχαριστώ όλους. Είναι τιμή μου να ομιλώ ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακόμα μια φορά. Κοιτώ γύρω μου, σε αυτή την ιστορική αίθουσα και βλέπω εκατοντάδες ανθρώπων. Στην πραγματικότητα όμως ε, είναι μαζί μας σήμερα πολλά εκατομμύρια επιπλέον από διαφορετικές χώρες, ιστορίες και προοπτικές. Εμείς που μαζευτήκαμε σήμερα εδώ